Welcome everybody. Καλώς όλοι. Καλώς ήρθατε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της Μέσης Διάταξης, πόλεμος στη Συρία, τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις και μελλοντικές προοπτικές. Και τώρα θα μιλήσω τσεχικά. Παρακαλώ, βάλτε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι κάπως ε, ασυνήθιστα θέτοντας ένα ερώτημα. Οι εκθέσεις που έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα 13 Μαρτίου μιλούν για την πολιορκία του Αφρίν από τις τουρκικές δυνάμεις και έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ξεκινήσει αυτή η πολιορκία από ό,τι φαίνεται στο Αφρίν θα επαναληφθεί αυτό που συνέβη στην Ανατολική Γκούτα. Πρώτα βομβαρδισμός και τώρα ε, πολιορκία. Και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ε, πολίτες και στο Αφρίν όπως και στην Γκούτα. Και βεβαίως ε, αυτό το μπλόκο δεν επιτρέπει στην ανθρωπιστική βοήθεια να μπει στην πόλη. Εκατοντάδες πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν φάρμακα. Αλλά στην Κούτα είναι οι ρωσικές δυνάμεις και ο στρατός του Ασάντ. Στο Αφρίν όμως ε, οι Τούρκοι είναι αυτοί που βαρτίζουν Και θέλω το ερώτημα αυτό τώρα, πριν τη συζήτηση. Ο τουρκικός στρατός, ο οποίος σκοτώνει αθώους πολίτες, είναι σύμμαχος προς εμάς. Θα ήθελα να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και θα ήθελα να γίνει αναφορά στο τι συμβαίνει στο Αφρίν και για το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή ε, οι δυνάμεις που υποτίθενται είναι τουρκικές. Επτά χρόνια έχει κρατήσει αυτός ο πόλεμος και νομίζω ότι δεν μπορούμε απλά να συζητάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να βρούμε βεβαίως τρόπους και να συζητάμε θα δώσω, θα καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες εδώ, θα ήθελα να μας ενημερώσουν για τις εξελίξεις και την προοπτική του να εξευρεθεί κάποια λύση σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς τέλος. Να καλωσορίσω τον Jean-François ο οποίος είναι πολιτικός εξωματούχος για τη Συρία και εμπειρογνώμονας σε ζητήματα ασφάλειας. Καλωσορίζω και την κυρία Φλόρενς Κάουμπ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις Μελέτες Ασφάλειας και ο Έρβιν Βαν Βέν ερευνητής από το Κλίνγκενταλ ε, το Ινστιτούτο των Κατοχωρών το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων των Κατοχωρών δεν έχουμε πολύ χρόνο θα πρέπει 12 και μισή να έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκάου. Ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Βεβαίως δεν είναι ο λόγος που έρχομαι εδώ χαρμόσυνος. Ε, πριν από τέσσερα χρόνια είχα ξαναέρθει και πάλι για τον πόλεμο στη Συρία μιλούσαμε. Έκτοτε τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς οι Ευρωπαίοι μου θέσατε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Και ξέρω ότι για πολλούς από εσά ε, το λέτε και στο ψήφισμά σα την προηγούμενη εβδομάδα, ε, είναι σημαντικό το ερώτημα που θέσατε. Αλλά αυτό που αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης ε, ε, και αναφέρουν κάποιοι σχολιαστές, ότι ο πόλεμος σύντομα θα τελειώσει, είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ απολύτως και κάθετα. Θα σα εξηγήσω γιατί. Είναι πάντω επικίνδυνο να πέσουμε στην παγίδα αυτή τη αυτής Η παρουσίαση που έχω προετοιμάσει ε, θέτει το θέμα του τι θα γίνει εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, να πιστέψουμε δηλαδή ότι θα, θα τελειώσουν σύντομα, ε, θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος και δεν θα είναι πλέον δικό μας πρόβλημα. Η έχουμε τις εξελίξεις επιτόπου, όχι μόνο οι τουρκικές επιχειρήσεις, αλλά και οι ρωσικές, ε, ε, αυτές της Συριακής κυβέρνησης, το γεγονός ότι ο, ο ISIS δεν είναι πια στη Συρία, ε, είναι μόνο σε κάποιους θύλακες και όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα και διπραγματεύσεις επί ρωσική εποπτεία, στη τελευταία συνάντηση στο Σότσι επετεύθη μια συμφωνία βασική για να συζητηθεί ένα νέο σύνταγμα για τη Συρία, όλα αυτά δημιουργούν την ψευδέστηση ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Έχει περάσει και πολύ καιρό. Ε, πολλοί λοιπόν τους αρέσει να, σκεφτούν ότι αφού έχουν περάσει, να σκέφτονται ότι αφού έχουν περάσει 7, 7 χρόνια θα πει ότι είμαστε κοντά στο τέλος. Δυστυχώς εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αξιολόγηση και δεν συμφωνούν και πολλοί άνθρωποι ε, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή και θα ξέρουν κάτι περισσότερο για τους λόγους αυτής της σύραξης ε, περισσότερο από εμά. Το τέλος του πολέμου στη Συρία δεν είναι το τέλος ε, της, των σειράξεων στη Συρία. Τι θα πει αυτό. Η σύραξη ξεκίνησε λόγω, για κάποιους λόγους. Ο πόλεμος είναι μια έκφραση αυτής της σύραξης, αυτής της διένεξης. αν δεν εμπληθεί το πρόβλημα, ε, ε, ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος το 2011, η βία θα συνεχιστεί. Εντάξει, θα πάρει άλλους μορφές. Τώρα έχουμε ε, πόλεμο εδάφους, αλλά μπορεί να πάρει άλλες μορφές η βία. Στατιστικά στοιχεία εδώ μας λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής δεν πιστεύουν ότι θα τελειώσει αυτός ο, αυτός ο πόλεμος ούτε φέτος ούτε του χρόνου ούτε τα επόμενα πέντε χρόνια. Γιατί είναι τόσο απεσιόδοξοι, τι γνωρίζουν που δεν γνωρίζουμε εμείς. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Είναι η ρίζα του κακού, η ρίζα ε, της διένεξης αυτής. Δεν είναι ε, μόνο δική μου άποψη. Ξέρετε, μία διένεξη δεν φεύγει έτσι. Εάν δεν επιληθεί το πρόβλημα ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η διένεξη ε, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες βεβαίως που το υποστηρίζουν αυτό. Καταρχήν δεν έχει λήξει ο ίδιος ο πόλεμος. Επίσης, ε, κανείς στη Συρία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί στρατιωτικά να ελέγξει το σύνολο της χώρας. Το σύνολο, το σύνολο της χώρας. Η ασφάλεια λέει θα παραμείνει ως πρόβλημα. Άλλο είναι να κάνει κάποιος μια επίθεση να, και να ε, κατακτά εδάφη και ένα άλλο πράγμα είναι να σταθεροποιεί ε, την κατάσταση μετά. Άλλο να κερδίσει τον πόλεμο, άλλο να κερδίσει την ειρήνη. Σκεφτείτε τι έγινε στο 2011 ε, και, και, και μετά αλλού. Ε, οι αστυνομικέ δυνάμει τη Συρίας πάντως, αυτό που έχει μείνει από αυτέ, δεν μπορούν να εγγυηθούν ε, την ασφάλεια πέρα από κάποιε περιοχέ Και θα παραμείνουν περιοχέ ολόκληρε εκτό ελέγχου και ούτε η Ρωσία ούτε η Ιράν, το Ιράν θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές ως δυνάμεις ε, εγγύητρες στην περιοχή. Και βέβαια υπάρχουν και τα χρήματα. Υπάρχει μεγάλη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να, δώσουν, να δώσει χρήματα για την ανοικοδόμηση. Μιλάμε για 100 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση. Τεράστιο ποσό. Και βεβαίως τα χρήματα δεν λύνουν τα προβλήματα από μόνα τους δεν φτάνει μια πιστοτική κάρτα για να λύσουμε το πρόβλημα. Εφόσον η κατάσταση ε, δεν σταθεροποιηθεί σε επίπεδο ασφάλεια, ε, η ανοικοδόμηση δεν σημαίνει τίποτα. Είναι σαν να γεμίζουμε ένα βαρέλι χωρί πάτο. Και η χρηματοδότηση δεν λύνει τα, προβλήματα. Θα υπάρχει ανασφάλεια, δεν θα υπάρχει απασχόληση. Θα είναι ένα μη σταθερό περιβάλλον, εν περιπτώσει. Είπα ότι το πιο βασικό είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη ρίζα του κακού. Στη Δαμασκό αυτή τη στιγμή, λόγω της, ε, των νικών ε, στον πόλεμο, δίνεται η εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να κάνουν υποχωρήσεις και δεν κάνουν υποχωρήσεις, δεν κάνουν ε, Λαμβάνω χώρα διαπραγματεύσει λοιπόν στο Σότσι, αλλά ο νέο οδικό χάρτη για, για το νέο Σύνταγμα δεν τη χάνει υποστηρίξει από διάφορου εμπλεκόμενου. Είμαστε ακόμα σε μια πολύ βίαιη φάση. Τι σημαίνει αυτό για μα, Πρώτα απ' όλα έχουμε επίπεδα βίας ε, ε, ανταρτοπολέμου στη Δαμασκό ε, αλλά και αλλού στη χώρα, ίσω ε, τα πράγματα εξελιχθούν όπω το Ιράκ να στο 2004 και το 2008. Επίπεδο λοιπόν βία το, το οποίο είναι αρκετό για να μην επιτρέπει καμία πολιτική μεταρρύθμιση και ούτε και κάποια οικονομική δραστηριότητα. Ούτε, ούτε η Ρωσία ούτε το Ιράν είναι σε θέση οικονομικά ή πολιτικά να ε, μπορέσουν να παραμείνουν στη χώρα. Είναι όπω οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, στο Ιράκ μετά το 2004. Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν δηλαδή την σταθεροποίηση. Είναι κάπως κοινικό αυτό αλλά ε, το γεγονός ότι θα συνεχιστεί ακόμα λίγο η σύραξη σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές κάποια στιγμή θα φτάσουν στα όρια τους και θα κάνουν κάποιες παραχωρήσεις, θα κάνουν τις απαραίτητες παραχωρήσεις για να φτάσουν σε συμφωνία. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό άμεσα. Αυτό για μας, κυρίως για τις χώρες στην περιοχή μάλλον, ε, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πιο πολλοί πρόσφυγες, δεν θα επιστρέψουν στη Συρία οι πρόσφυγες, ε, δεν θα είναι ασφαλής η κατάσταση για να επιστρέψουν και τέλος, ε, είναι κάτι ξεχωριστό βέβαια, πρέπει να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αν θεωρείτε ότι ο Άισις ε, τελείωσε, δεν θα συμβεί αυτό, θα επανέλθει από άλλη μορφή. Και η Αλκάιντα είναι ακόμα ενεργή και στη Συρία. Αυτό το πολιτικό κενό λοιπόν που υπάρχει στη Συρία θα οδηγήσει στο να εμφανιστούν νέοι τζιχαντιστές και θα βρεθούμε εκεί που βρισκόμασταν πριν από 7 χρόνια. Τα αναφέρω όλα αυτά, ε, τα οποία τα ξέρετε φαντάζομαι, διότι γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ε, η φωνή του ακούγεται, ο ρόλος σας να συνεχίζεται να παραμένει ανοιχτή αυτή η πληγή, να μην, δοθ, να μην περάσει ότι όλα θα πάνε καλά με τους Ρώσους και τους Σύριους και τους Ιρανούς. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος βιώσιμα είναι να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Σημαίνει δηλαδή σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και βεβαίως μια κυβέρνηση που να λογοδοτεί, διότι εκεί ξεκίνησαν όλα πριν από 7 χρόνια. Αυτή η φωτογραφία ε, την είχα πάρει το 2010. Δεν ξέρω τι έγινε με τα παιδιά αυτά έξωτε, αλλά για αυτούς τελικά, για αυτά τα παιδιά τελικά, θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια, να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει άλλη λύση σήμερα στη Συρία από το να λάβουν χώρα αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και απλό, αλλά είναι σημαντικό. Σα ευχαριστούμε, Νομίζω πως ε, αυτή η οπτική γωνία του να μην είμαστε υπερβολικά αισιοδοξοί ενδεχομένως θα μας οδηγήσει σε περισσότερα αποτελέσματα. Αλλά το λόγο δίνω τώρα στον Ζαν Φρανσουά ε, για την παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρουσίαση της κατάστασης της Συρίας και το τι μπορούμε να δούμε και να πω ότι συμφωνώ με κάτι που είπατε εσείς και θα μπορούσα να το είχα πει και εγώ. Αλλά ίσως κάποιος, κάπως πιο αδέξε και όχι τόσο κομψά όπως το είπατε εσείς. Συμφωνώ λοιπόν σε σχέση με το σχόλιο που κάνατε ότι η σύραξη δεν έχει φτάσει στο τέλος της. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη στρατιωτική στη Συρία. Ακόμα δηλαδή και αν ε, το καθεστώ του Ασάντε και οι σύμμαχοί του ε, εδώ και ένα, ενάμιση χρόνο έχουν καταφέρει κάποιες σημαντικές νίκες, η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Γιατί θα, η, ε, ο ρόλος των τρομοκρατικών ομάδων ε, και του Ισλαμικού κράτους θα διαφοροποιηθεί. Θα ξεκινήσω καταρχήν από την κατάσταση, με την κατάσταση στη Δαμασκό και στην Ανατολική Κούτα γιατί εκεί η κατάσταση και στο Αφρίν είναι ακριβώς τα δύο ε, ζητήματα που μας ανησυχούν περισσότερα από τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε ότι εδώ και παραπάνω από ένα μήνα ε, το καθεστώς Ασάτ και οι σύμμαχοί του ξεκίνησαν μια επίθεση κατά της Βούτα, ε, ξεκίνησε με μια αερια επίθεση, δηλαδή με βομβαρδισμούς εναέριους και στη συνέχεια ακολούθησε χερσαία επιδρομή από τις από, το, από τις ε, χερσαίες ε, δυνάμεις, από τις ε, κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά και παραστρατιωτικές δυνάμεις. Και ε, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 60 με 70% της Ανατολικής Κούτα, χρησιμοποιώντας ό,τι μπορούν να κάνουν, δηλαδή βομβαρδισμούς και με αέριο χλωρίνης και με α, βομβαρδισμό και των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και επιθέσεις κατά αμάχων. ο φόρος αίματος ε, για αυτή την επίθεση στην Ανατολική Γκούτα είναι 1.400 άμαχοι νεκροί μέχρι στιγμής. Τώρα, ε, στα νότια προάστια της ε, Δαμασκού, αναφέρατε ότι υπάρχει εκείνη ένας μικρός θύλακας υπό τον έλεγχο ακόμα του ISIS και πριν από μερικές μέρες είδαμε κάποιες συγκρούσεις μεταξύ του ΑΣΥΣΕ και των ε, Συριακών Κυβερνητικών Δυνάμεων. Τώρα, εάν πάμε λίγο ε, προς τα βόρεια και την ε, κοινή επιχείρηση εκεί των τουρκικών δυνάμεων και των συμμαχικών δυνάμεων της Συρίας, θα δούμε ότι ξεκίνησε και αυτή η επιχείρηση πριν από ένα μήνα η α, τουρκική πλευρά κατάφερε να θέσει από τον έλεγχό της ένα σημαντικό τμήμα αυτής της ε, περιοχής και ο στόχος της Τουρκίας, τουλάχιστον αυτό λέει, είναι ότι θέλει να καταστήσει ασφαλή τα σύνορά της με τη Συρία και γι' αυτό είναι διατεθειμένη να κινηθεί και πιο πολύ προς τα ανατολικά, δηλαδή προς τα σύνορα με το Ιράκ. Αλλά αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα από την Τουρκία είναι να ε, ε, καταλαβαίνει τον έλεγχο του Αφρίν μέσα σε ένα μήνα. Από, ξεκινώντας δηλαδή από τα σύνορα βρέθηκα ειρήνη στο Αφρίν. Και αυτό που ε, διαπιστώνουμε είναι ότι οι συμμαχικές ε, δυνάμεις μετά από αυτήν την ε, δρομή δεν κάλεσαν τον πληθυσμό να επιστρέψει στις αιτίες του. Οπότε φοβούμαστε ότι γίνεται μια προσπάθεια μετακίνησης πληθυσμών, δηλαδή να εκδιωχθούν όλοι οι Κούρδοι από το Αφρίν και να επανεκατασταθούν άλλοι ε, ε, πληθυσμοί εκεί. Δηλαδή αντίστοιχο ακριβώς με αυτό που είδαμε στη Ράκα. Τώρα από εκεί και μετά υπάρχουν ε, άλλα ζητήματα σειράξης στην ίδια τη Συρία. Καταρχήν ο πόλεμος κατά του ISIS, ουσιαστικά το SDF και η Παγκόσμια Συμμαχία κατά του ΝΤΑΕΣ κατάφερε να περιορίσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό ε, την, ε, το ISIS, ε, καταλήφθηκε η Ράκα πέρυσι, τώρα κατάφερα να ελέγξουν και τα σύνορα και ουσιαστικά όλες οι επιχειρήσεις που συνεχίζονται σε αυτή την περιοχή στοχεύουν ακριβώς στο να εξαλειφθεί πλήρως η παρουσία του ISIS στα νότια του, της χιλάδας του Εφράτη και στα σύνορα με το Βόρειο Τώρα, σε ό,τι αφορά το νότο της χώρας, ε, ε, ε, αυτή είναι η περιοχή δηλαδή την οποία ονομάζουμε ως περιοχή αποκλιμάκωσης ουσιαστικά σε δύο τμήματα αυτής της περιοχής ουσιαστικά έχουμε κλιμάκωση αντί για αποκλιμάκωση. Τώρα, στα νότιο-δυτικά, όπου είχαμε να κάνουμε μια σχετικά ήπια περιοχή, αν μπορούμε να την κατονομάσουμε ως τέτοια, υπήρξαν κάποιοι μοβαρδισμοί από το Συριακό καθεστώ τη. αλλά αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι γίνονται κάποιε διαπραγματεύσει μεταξύ του καθεστώτο Ασάτ και ε, του ε, οι οποίε όμω ακόμα δεν έχουν προχωρήσει αρκετά. Και η τελευταία μεγάλη περιοχή η οποία μα ενδιαφέρει βέβαια είναι το Ιντλίπ. Ε, συνεχίζεται καταρχήν η σύραξη ε, μεταξύ των ε, απονεμαριών ή μάλλον μεταξύ Αλσάμ και Αλζίνκη και ε, των υπολοιμάτων της Αλκαΐδα και του μετώπου Αλνούστρα. Ουσιαστικά η Αλκαΐδα έχει υποχωρήσει από αυτήν την συμμαχία η οποία λαμβάνει και την υποστήριξη της Τουρκίας αλλά βλέπουμε πως υπάρχει ταυτόχρονα και σύραξη μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και αντιφρονούντων στα νότια της ε, περιοχής του Ιντλίπ. Τώρα, αν θέλουμε λίγο να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές. Αυτό που παρατηρούμε κατά τους ε, τελευταίους ε, μήνες είναι από τη μία πλευρά το πεδίο μάχης να καθίσταται πιο περίπλοκο, αλλά από την άλλη πλευρά να γίνεται πιο απλό. Ε, δηλαδή, ε, μέχρι τα τέλη του έτους μπορεί να έχουμε τέσσερις μεγάλες ε, περιοχές στη Συρία. Καταρχήν θα έχουμε την περιοχή που θα ελέγχεται από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Μετά, ε, τις εκτεταμένες ε, βορειο περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους. Μετά, οι περιοχές της ε, τουρκικής παρέμβασης, και εδώ αναφέρομαι στην επιχείρηση Shield στον Ευφράτη και στην επιχείρηση Olive Branch αλλά και στην, ε, στις περιοχές, ε, στο μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής Idlib η οποία θα ελέγχεται όπως είπαμε από αυτές τις συμμαχιές δυνάμεις που τον έχουν της Τουρκίας και μετά τέλος η τέταρτη περιοχή θα είναι η νότιο-δυτική όπου ε, θεωρούμε πως στην πραγματικότητα θα συνεχίσει να υποχωρεί το ISIS αλλά θα αρχίσει να προσαρμόζει ε, και να κινείται πιο πολύ προς τον άνταρτο πόλεμο όπως το κάνει ήδη σε ορισμένα τμήματα της Συρίας. Και πράγματι δεν έχουμε δει ε, σημαντικές ενέργειες του ISIS ε, το τελευταίο καιρό. Βέβαια τα όσα συνέβησαν στο Αφρίν δεν βοηθάει το ασες ε, γιατί το ΕΣΤΕΝΕ και το PID ε, βρέθηκαν στην εχμή αυτής της επίθεσης ε, που χρειάστηκε ότι χρειάστηκε να αποσπαστούν κάποιες από τις δυνάμεις τους από εκείνη την περιοχή στο Αφρίν. Κάτι τέτοιο βέβαια έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την επιχείρηση της Παγκόσμιας Συμμαχίας. Θα σταματήσω εδώ και είμαι βέβαια στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήματα. Ευχαριστούμε, Ζαν Φρανσουά. Το λόγο έχει τώρα ο Έρβιν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Κύριε Πρόεδρε, θα προσθέσω και δυο σκέψεις στα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Θα ξεκινήσω λίγο προκλητικά και θα το αναπτύξω ως επιχειρηματολογία στη συνέχεια. Μπορούμε να πούμε ότι η αρχική σύγκρουση έχει τελειώσει. Την κέρδισε ο πρόεδρος Ασάντ και οι διεθνείς του σύμμαχοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο πόλεμος. Διότι ε, είδαμε τι είπε η κυρία Γκάουμπ, είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ο, τον πόλεμο τον κέρδισε το αυταρχικό καθεστώς. Οι δύο παραγόντες που θα καθορίσουν και θα επηρεάσουν σημαντικά τη διάρκεια της σύραξης αυτής, της σύγκρουσης αυτής, θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα καταλήξει συμφωνία με τις κουρδικές δυνάμεις ε, η κυβέρνηση και κατά πόσο θα συνεχίσει να υποφελείται από αμερικανική στήριξη στα ανατολικά της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να έχουμε πολιτική μετάβαση βραχυπρόθεσμα ούτε μεσοπρόθεσμα. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν έχει τέτοιο πολιτικό ενδιαφέρον το καθεστώς. Ε, θα κάνει ίσως κάποια δίθεν μετάβαση, δημιουργώντας κάποιες ε, δίθεν αντιπολιτευτικές ομάδες ε, που θα συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι να γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η ανοικοδόμηση, υπό τους όρους της κυβέρνησης φυσικά. Βασίζεται σε, εστιάζεται σε αστικές περιοχές, κλειδί στη Δαμασκό κτλ. Θα το δούμε αργότερα με λεπτομέρειες. Το άλλο πρέπει να αναρωτηθούμε είναι σε ποιο βαθμό αυτό καθιστά τι δυτικέ διαπραγματευτικέ πολιτικέ στη διαδικασία της Γενέβη, ε, το να προστατεύουμε τους πρόσφυγες ε, εφικτές. Και τέλος, το Ισλαμικό κράτος προφανώς δεν έχει ιτηθεί. Οι αιτίε που οδήγησαν στη γέννησή του, τα οικονομικά του δίκτυα, οι πόροι του, απλά έχουν περάσει στην απόλυτη, έχουν γίνει απολύτως αόρατα. Και ξέρουμε ότι πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τη Συρία και πολλές τέτοιες οικονομικές κινήσεις. πολλέ πολλές από αυτές που αποτελούσαν γραμμή ζωής για πολλούς ε, Σύριους και Ιρακινούς. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Δύο σκέψεις για τη φύση του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Θα μας βοηθήσει αυτό να καταλάβουμε τι μορφή θα έχει οποιαδήποτε ανοικοδόμηση. Και μετά θα τελειώσουμε κάποιες σκέψεις για το τι θα μπορούσε να γίνει στη θέση όλων αυτών. Μετά από την τελευταία, ε, τελευταία επταετία παρατηρούμε ότι η σύγκρουση αυτή μεταμορφώθηκε με διάφορους τρόπους από διαμαρτυρία σε ανταρσία, σε πόλεμος και σε κάποια μορφή, κάποια μορφή σταθεροποίησης ε, που βλέπουμε τώρα. Το αποτέλεσμα είναι ε, πολλά διαφορετικά συμφέροντα σε ένα συγκεκριμένο χώρο χωρίς να έχουν το ίδιο βάρος όλοι. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η σύγκρουση χαρακτηρίστηκε από τη σύγκρουση τόσων πολλών συμφερόντων που είναι πολύ δύσκολο να τα διαχωρίσουμε. Όταν μιλάμε για ανοικοδόμηση λοιπόν ε, για την κλασική προσέγγιση της ανοικοδόμησης μέσω μιας συνθήκης ειρηνευτικής ε, ε, όλο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση. Όπως είπε η κυρία Γκάουπ, η βία μπορεί να μειωθεί σε ένταση, έχει ήδη μειωθεί σε πολλά μέρη, αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο, διότι οι αιτίες ε, της ε, αβεβαιότητας υπάρχουν ακόμα και ενισχύονται όσο πιο πολύ εγκαθιδρύεται ισχυρά το αυταρχικό καθεστώς του Πρόεδρου Ασάντ. Τι σημαίνει αυτό για την ανοικοδόμηση που αρχίζει να εμφανίζεται αργά-αργά στις πολιτικές συζητήσεις, στον ορίζοντα. Συγκρίνοντας με άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε ότι το χρήμα δεν αγοράζει την αγάπη. Με άλλα λόγια, όσα και να επενδύσει κανείς, δεν πρόκειται να επιτύχει τις πολιτικές παραχωρήσεις σε ζητήματα προσφυλή στην κυβέρνηση. Οπότε αυτό το σκεπτικό πρέπει να το απορρίψουμε, διότι υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να γίνει η ανικοδόμηση θα αντιστοιχεί στη λογική μάχης ε, του καθεστώτος. Δηλαδή θα τιμωρηθούν όσοι ήταν αντίθετοι στο καθεστώς, θα σκεφτεί το καθεστώς ποια είναι η βάση του και αυτήν θα υπερασπίσει. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ανικοδόμηση θα είναι ε, σταδιακή, επιλεκτική, θα υποφελεί τις ομάδες και τις περιοχές ε, που υποστήριζαν το καθεστώ. Οπότε το καθεστώ δεν πρόκειται να βιαστεί να επαναφέρει τους πρόσφυγες που έφυγαν στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Αυτό που θα δούμε μάλλον θα είναι την επανεγκατάσταση του αυταρχισμού. Μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται σε ολόκληρη τη Μέση Και αυτό γεννά διάφορα ερωτήματα. Όταν μιλάμε για γνήσια πολιτική μεταρρύθμιση, όπως λέτε εσείς ε, σε διάφορα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρόσφατο ψήφισμα, προβλέπουμε έλλειψη λογοδοσίας μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και φυσικά το βασικότερο πρόβλημα στην περιοχή θα είναι ότι οτιδήποτε γίνει θα είναι απολύτως μη βιώσιμο. Δύο πράγματα πριν κλείσω, διότι όλα αυτά εντάξει τα λέμε εμένα, αλλά ποια είναι η εναλλακτική. Δεν φαίνεται να υπάρχει ενδεχόμενο στρατιωτική ε, επέμβαση αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τι Αμερικανικέ δυνάμει που είναι παρούσε Έχω να πω τρία πράγματα. θα πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τη ε, διασπορά από τη Συρία. Έχει έρθει για να μείνει, θα μοιάζει με την Παλαιστινιακή διασπορά του 20ου αιώνα. Πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το καταπληκτικό δυναμικό να αποκτήσουν θεσμική εμπειρία, δημοκρατική εμπειρία, ώστε οι μνήμες αυτές να μείνουν ζωντανές στα μυαλά τους όταν θα έρθει η στιγμή που θα μπορέσουν να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν στη χώρα τους. Δεύτερον, το Ιράν θα πρέπει να συμμετέχει πιο οργανωμένα και αυτό να προκληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα του Ιράν στη Μέση Ανατολή είναι σημαντικά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε μαζί τους, αλλά θα πρέπει να τους έχουμε ως ισότιμους συμμετέχοντες ε, και μιλώντας ανοιχτά, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή επαρκώς. Και τέλος, πάμε να θυμηθούμε τη δεκαετία των 90. Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση σε κάποιο βαθμό στα Βαλκάνια, όπου για πολλά χρόνια είχε διαδοθεί το οργανωμένο έγκλημα, η ριζοσπαστικοποίηση, πολλά αρνητικά, πολλές αρνητικές συνέπειες που μπορεί να βλέπουμε στο μέλλον από τη Συρία και τον πρόεδρο Ασάντ και που μπορεί να ενταθούν. Ποια στρατηγική λοιπόν θα βοηθήσει να διατηρήσουμε την περιοχή ασφαλή από διάφορες απειλές που μπορεί να προκύψουν από τη Συρία και να διατηρήσουμε ασφαλείς και τους εαυτούς μας, εάν οι σημερινές εξελίξεις πολλαπλασιαστούν ε, ως συνέπεια στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ας ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα. Θα ήθελα να ε, παρακαλέσω τους ομιλητές να περιοριστούν ε, στο 1,5 λεπτό ώστε να έχουμε και χρόνο να απαντήσουν τα μέλη του πάνελ. Ε, πρώτη κυρία Λέζιν. Ja, Σας ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με το ερώτημα που έθεσε ο Πρόεδρος και θα ήθελα να το συμπληρώσω ως προ την οπτική γωνία την εξή. Και εδώ απευθύνομαι κυρίως στον κύριο Βανφέν. Ε, πώς βλέπετε, πώς αξιολογείτε την τουρκική παρέμβαση στο Αφρίν με βάση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Και σε εσά, ε, κυρία μου, να σας ρωτήσω ε, ποια θα θεωρούσατε πως είναι η κατάλληλη δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα μετά από τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν ότι προτίθεται να συνεχίσει αυτή την στρατιωτική επίθεση. Και από εκεί και μετά, από ό,τι διάβασα στη Λιβανέζικη εφημερίδα Αλαπά, υπάρχει ένα πρωτόκολλο ε, το οποίο δημοσιεύθηκε από συνάντηση μιας μικρής ε, ε, ομάδας στην πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου ε, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά την κατανομή της Συρίας, το διαμερισμό της Συρίας. Γνωρίζετε εσείς κάτι ε, σχετικό με αυτό. Υπήρχε μια τέτοια συζήτηση και αν πραγματικά έλαβε χώρα μια τέτοια ε, συζήτηση, ποια είναι τα συμπεράσματα που αντλεί είπατε εκπρόσωπος για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την αδερφική ακαιρεότητα και το αδιέρωτο της Συρία. Ευχαριστώ κύριε σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από αυτή την εξαιρετική παρουσίαση των τριών ομιλητών μας, ε, είναι δύσκολο να θέσει κανείς ένα εύστοχο ερώτημα, αλλά κυρία Λόζινγκ ε, τα κατάφερα να θέσει πολύ εύστοχα ερωτήματα, οπότε θα πρέπει και εγώ από τη ε, σειρά μου να θέσω κάτι αντίστοιχο ως ερώτημα. Ένα λοιπόν ζήτημα που με απασχολεί από τότε που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου είναι το, το τι θα συνέβαινε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διέχεται μια ισχυρή, σταθερή, στεβαρή εξωτερική νη πολιτική. Ε, και για παράδειγμα υπήρχε εδώ και 7 χρόνια. Ε, νομίζω πως αν είχαμε τότε δηλαδή στην ε, έναρξη της σύραξης μιλήσει με ένα, ένα φωνή, ένα ενιαίο μέτωπο, και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν συνέβη σε άλλες περιοχές και το τι μπορεί να επιτευχθεί με τη διπλωματία, μήπως θα είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις μικροσυράξεις που είχαν ξεκινήσει. Προκειμένου δηλαδή να μην ε, εξελιχθούν αυτές οι ε, εμπόλεμη σύραξη. Μήπως θα μπορούσαμε δηλαδή ε, να έχουμε βοηθήσει τις διάφορες πλευρές να αποφύγουν αυτό το μεγάλο πόλεμο που ξεκίνησε. Γιατί γνωρίζουμε ε, πως οι συνέπειες αυτού, ε, αυτού του πολέμου έχουν πλέον φτάσει και στις δικές μας χώρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις άριστες παρουσιάσεις. Ναι, αυτές οι περιοχές κλιμάκωσης, όπως είπατε, είναι μέρη που κατακρεματίζουν τη χώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση είναι κατά την άποψή σας θα σταθεροποιηθούν θα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο κάποια επίσημη αναγνώριση των διαφόρων δυνάμεων, των διαφόρων εξι... ισορροπιών ε, εξουσίας. Δεύτερη ερώτηση, πώς θα επιδράσει τη σύγκρουση, η πιθανή αμφισβήτηση από τον πρόεδρο Τραμπ της συμφωνίας με το Ιράν. Η διαφορετική αυτή στάση που θα μπορούσε να αναμένει κανείς και από, τους δύο, από τις δύο πλευρές ε, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Προτελευταία ερώτηση όσον αφορά την κατάληψη του Αφρίν ε, και τις δράσεις της ε, τουρκικής κυβέρνησης που φιλοδοξεί να επεκταθεί. Έχει το στόχο να φτάσει στο Ακομπάν. Κατά την άποψή σας, πώς ε, θα επηρεάσει αυτή η τουρκική εισβολή τους πιο σημαντικούς παίκτες του σύγκρουσης, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, δεδομένου ότι η Ρωσία φαίνεται να το έχει δεχτεί. Και τι τριβές θα δημιουργήσει με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κόουσο. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ διαφωνώ με κάποια ζητήματα που ακούστηκαν. Ε, καταρχήν δεν συμφωνώ με κανέναν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα αρχέτυπο ε, εμφύλιο πολέμου ε, μάλλον μοιάζει με τους καινούριου πολέμους. Ε, πολλαπλασιασμός των εμπλεκομένων, ε, κατακαιρματισμός, ε, ασύμετρες μέθοδοι ε, μάχης, τρομοκρατία, ε, χρήση βίας, βαρβαρότητες είναι όπως κατά κάποιο τρόπο με, το, με την ε, Αραβική Άνοιξη. Ε, ήδη το 1973, το 82, ε, οι αδερφοί μουσουλμάνοι είχαν προετοιμάσει, είχαν, είχαν κάνει εξεγέρσεις. Το 73, σας θυμίζω, για μια αλλαγή ε, στο Σύνταγμα όπου είχε δοθεί ε, μια θέση ε, επικεφαλής μουσουλμάνου αλλά ήθελαν να είναι Σουνίτης τότε οι αδερφοί μουσουλμάνοι το 1973. Ε, ξέρετε, η ελεύθερος στρατός της Συρίας τελικά διαλύθηκε και πήρε τη θέση του η Αλκάιδα και ο Άισις και τελειώνω πρόεδρε. Ούτε με τη Λιβύη μπορούμε να συγκρίνουμε στην Κούτα, στην Ανατολική Κούτα έχουν τελειώσει τα πράγματα. 90%. 90% έχει καταληφθεί. και οι τρομοκράτες φεύγουν προς το Ιντλίμπ. Εκεί είναι και η Αλκάιντα, είναι το Αλ-Ισλάμ που επιτίθενται, επιτίθενται με όλμους εδώ και μέρες, με δύο νεκρούς ήδη σήμερα, πάνω από 200 τελευταίες μέρες. Και τι θα γίνει με την Τουρκία βέβαια, που ε, αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει το, τη Συρία, Συρία, το Συριακό στρατό το Τεν Αλτζαμπίν. Ο Γιούρεκ έχει το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα γενικό ερώτημα. Δεν ξέρω αν πρέπει να επικεντρωθούμε στο να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε τη δημιουργία μιας διεθνούς προσέγγισης. Εδώ και χρόνια κρατάμε φίλος πόλεμος, προσπαθούμε να, να δούμε ποιος θέλουμε να κερδίσει καταρχήν. Ε, στη Συρία για χρόνια είχαμε ένα γεωπολιτικό πρόβλημα. Ήταν μια απειλή προς τους νότιους γείτονες αυτή είναι η βασική πρόκληση ε, τη, της πολιτικής ε, του καθόλου του Ασάντα. Και υπάρχει ένα θέμα ανοχής βέβαια στο εσωτερικό επίπεδο. Αν και δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όπως παραδείγματος χάρη στη Σαουδική Αραβία σε ό,τι φορά τον αυταρχισμό. Εδώ όμως υπάρχει ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Θέλουμε να μειώσουμε τον ανθρώπινο πόνο και να αποφύγουμε την κλιμάκωση. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν. Η ασφάλεια των γειτονικών χωρών δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και στη Συρία. Ίσως να πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια ε, ρεαλιστική λύση έτσι ώστε η Συρία να είναι μια χώρα που να είναι λιγότερο απειλητική για το διεθνές, την διεθνή τάξη πραγμάτων. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Δεν ξέρω, μπορεί να μου διέφυγε. Δεν μάθαμε τι έγινε με την αποστολή του Στέφαν Ντεμίστερα. Επίσης με την Κούτα Ποιος είναι εκεί στην Κούτα, μιλάμε για πολίτες, ε, άμαχο πληθυσμό, γιατί υπάρχουν και ομάδες ε, που έχουν πολιτικές ε, έτσι, προτιμήσεις. Ευχαριστώ κύριε Γιούρεκ. Λοιπόν, είχαμε πέντε παρεμβάσεις, τώρα έχουμε τρεις ομιλητές για να απαντήσουν και έχουν πια έξι λεπτά. Οπότε ο καθένας από εσά έχει δύο λεπτά για να απαντήσει. Ναι, ευχαριστώ. Ακούστε για να συνοψίσω λίγο και τα ερωτήματά σας. Πρώτον, η θλιβερή αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν είναι καλός στην επίλυση ε, σειράξεων. Ε, δεν νομίζω να είναι θέμα δράσης. Ε, από ό,τι φαίνεται όλο και πιο πολύ κρατώνει οι φίλοι πολέμοι. μετά το, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο μάλλον, έχουν, έχουμε όλο και πιο πολλούς ε, τοπικού ε, φίλους πολέμου ούτε εμεί δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί κρατάνε τόσο πολύ. Για την ερώτηση τη κύρια κυρίας, Λούζινγκ, ε, έχει σωστέ ιδέε ε, η Ευρώπη για το πώς να λύσει το πρόβλημα. Το θέμα, και εδώ επανέρχομαι και με τον κύριο Φρόιντ, είναι πώ επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι, ενώ έχουμε μία οντότητα η οποία ακολουθεί το δίκαιο ε, από τη φύση της. Ε, και είμαστε σε μια περιοχή που κανείς δεν ακολουθεί το δίκαιο. Οπότε οι Ρώσοι, οι Ιρανοί, οι διάφοροι, οι Τούρκοι, ακόμα και οι Αμερικανοί είναι μπροστά από εμά. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι μόνο θέμα να σχολιάσουμε την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλεία, είναι και το τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μα για να πετύχουμε του στόχου μα. Από την αρχή είχαμε πει ότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στη Συρία ε, είναι σωστό, αλλά δεν το υποστηρίξαμε με τα κατάλληλα μέσα. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία θα πρέπει να έχετε εσείς, να κάνετε εσείς και με άλλους πολιτικούς θύνοντες βεβαίως Ευρωπαϊ, Ευρωπαίους. Αλλά όταν είναι αναγκαίο πρέπει να έχουμε κατά νου και την ε, χρήση της ισχύω. revenir sur le risque de partition de la ναι, θέλω να επανέλθω στο, σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο ε, απόσχησης της Συρίας. Ε, ναι, υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον πίνακα που δείξατε ε, με τα ποσοστά ε, για το πόσο καιρό θα μπορούσε να κρατήσει αυτό ο πόλεμο, πόσο εκτιμούμε ότι θα κρατήσει, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αυτό ο κίνδυνο απόσχηση ε, έχει να κάνει με το γεγονό ότι το καθεστώ είναι σε μια στρατιωτική λογική αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη λογική την έχει ε, επιβάλλει ε, την σύραξη. Δεν θέλει το καθεστώς να μπει σε μια διαπραγμάτευση συμπεριληπτική. Ε, σε μια πραγματική διαπραγμάτευση δηλαδή. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να οθήσουμε το σύνολο των συνομιλητών μας να πείσουν το καθεστώ να πάει στη Γενέβη στις των διαπραγματεύσεων. Διότι μόνο με διαπραγματεύσεων θα βγούμε από αυτήν την ε, διένεξη και μόνο μέσω μια πολιτική συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει όλου. Η, η στρατιωτική λογική τη Δαμασκού αυτή τη στιγμή εναντιώνεται ε, σε οποιαδήποτε επίλυση του ζητήματο τη Συρίας. Προ τα εκεί λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε και εμεί υποστηρίζουμε ε, την δράση του Στεφάν Ντεμιστούρα διότι οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία θα πρέπει να γίνει στη Γενέβη με βάση ε, την, το ψήφισμα 2254 διότι πρόκειται για ψηφίσματα και για συμφωνίες ισορροπημένες σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση, σε ό,τι αφορά τους στόχους, στόχοι οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί, πραγματοποιήσιμοι, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Δαμασκός ε, να αποδεχτεί να έρθει στο τραπέζι των πραγματεύσεων. Αυτά. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ δύο σύντομα σχόλια. Ε, ευχαριστούμε και για τα ερωτήματα. Το πού ξεκινάει η επίλυση της Συριακής σύγκρουσης. Ε, θέλουν βεβαίως να ελέγξουν εδαφικά τη Συρία ε, του καθεστώς του Δαμασκού να φτάσει στα σύνορα του 2011 και να ελέγχει πραγματικά την περιοχή. Τι συμβαίνει λοιπόν. Έχουμε τη Ρωσία και το Ιράν. Διότι χωρί τη Ρωσία και το Ιράν θα είχε λήξει για αυτή η σύγκρουση. Είτε θα είχε καταρρεύσει η Συριακή οικονομία, είτε οι δυνατότητε ε, ε, οι στρατιωτικέ του Συριακού στρατού δεν θα ήταν επαρκεί. Θέλουν όμω διαφορετικά πράγματα αυτέ οι χώρε. Η Ρωσία θέλει έναν, ισχυρό κράτο, ένα αξιόπιστο σύμμαχο. Το Ιράν δεν θέλει αυτό. Θέλει ένα πιο ε, αδύναμο κράτος και να υπάρχουν διάφορες οργανώσεις παραστρατιωτικέ, ε, ε, όπως ε, και στο Λίβανο, στο Ιράκ και στην ίδια χώρα. και είναι πολύ προβλέψιμο αυτό από το ρωσικό μοντέλο. Για να απαντήσω το ερώτημα λοιπόν στο Ιράν την περιφερειακή ασφάλεια θα πρέπει να υπάρξει κάποια έστω και άτυπη συμφωνία με το Ιράν για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα παράλληλα δίκτυα και δυνατότητε, διότι ήδη στον ορίζοντα ε, πριν από μερικές εβδομάδες βλέπουμε τα προβλήματα με την κατάρριψη του Ισραηλινού αεροσκάφους, ε, του πολεμικού αεροσκάφους. Οι Τούρκοι επιτίθενται στο Αφρίν διότι τους άφησαν οι Ρώσοι. Ε, Τώρα υπάρχει μια ενδεχόμενη συνα... συναλλαγή με τη Ρωσία για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ε, ε, και κάπου αλλού η Ρωσία να προσπάσει κάτι άλλο. Αυτή τη σκέψη ήθελα να πω τελευταία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ. Ήταν εξαιρετικές ε, οι παρουσιάσει μας έδωσαν πολλά νέα στοιχεία, ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω ότι θα ρωτήσω κι εγώ το εξή. Ο τουρκικό στρατός ε, που σκοτώνει άμαχους είναι σύμμαχό μας. Δεν βλέπω να έκανε κανεί την ερώτηση, πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί απάντηση. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες Τετάρτη 20, 25 Απριλίου πρωί και απόγευμα και την Πέμπτη 26 Απριλίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους Ερμηνείς και τα μέλη της Γραμματείας. Ευχαριστώ.